Έχουμε τα χτεσινά πρακτικά, δεν ξέρω αν έχετε σχόλια. Η δική μας ε, συνειδρίαση της Ολομέλειας ξεκινάει, εγκρίνονται λοιπόν τα πρακτικά. Χτες λοιπόν